το τελικό σχέδιο ημερήσια διάταξη όπως το ενέκρινε η διάσκεψη των Προέδρων σύμφωνα με το άρθρο 141 σας έχει μοιραστεί. Δεν έχει ζητήσει κάποιο αλλαγή στην ημερήσια διάταξη της Δευτέρας. Οπότε περνάμε στην Τρίτη. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ζήτησε μία δήλωση από την Αντιπρόεδρο της Κομισιόν και τη εκπρόσωπο για την κατάσταση στην Γεωργία για το θέμα της επιλεκτικής δικαιοσύνης και το θέμα του DJ Γκουλάβα, το οποίο θα πρέπει να μπει με ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη το απόγευμα. Ο κύριος Κρίστιαν Πρέντα τώρα θα υποστηρίξει το αίτημα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ομάδα του ΕΛΚ θα ήθελε να συμπεριληφθεί αυτό το θέμα, δηλαδή η συζήτηση της Γεωργίας και της επιλεκτικής δικαιοσύνης ε, που εφαρμόζεται ως διαδικασία σε αυτήν την χώρα. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα πιστεύουμε. Θέλουμε να συζητήσουμε το ζήτημα της δικαιοσύνης και το συσχετισμό μεταξύ δικαστικού συστήματος και πολιτικού συστήματος στη Δημοκρατία της Γεωργίας. Ζητούμε από τους φιλελεύθερους και σοσιαλιστές συναδέλφους μας ευρωβουλευτές που πάντα είναι στεναροί υπέρμαχοι της ε, γεωργιανής κυβέρνησης να αντιληφθούν ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και ζητούμε να υπερψηφίσουν αυτό το αίτημα. Ιδιαίτερα στρέφομαι προς τους σοσιαλιστές συναδέλφους που στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζουν τον Πρωθυπουργό που είναι επίσης επικεφαλής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος ε, στην Ρουμανία και έχει καταδικαστεί από τη ρουμανική δικαιοσύνη. Καλή στιγμή θα ήταν να τον εγκαταλείψουν. In favor, please. Έχει υπέρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω ότι υποστηρίζω σε γενικές γραμμές όλες τις πρωτοβουλίες που στόχο έχουν να καταδικάσουν την επιλεκτική δικαιοσύνη. Αυτό το οποίο θα ήθελα θα ήταν ε, να σκεφτούμε και αυτά τα οποία είπε ο συνάδελφο ε, από το ΕΛΚ για την επιλεκτική ε, δικαιοσύνη όταν αυτή ασκείται εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραδείγματο χάρη την επιλεκτική δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Ε, για παράδειγμα την επιλεκτική δικαιοσύνη στη Γερμανία, στην επιλεκτική δικαιοσύνη στη Γαλλία. Όλα αυτά θα ήταν πολύ καλά για το κοινοβούλιο μας. Ευχαριστώ διακόπτη Πρόεδρος. Είναι κάποιος κατά παρακαλώ. Ο κύριος Γκερέρο. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική η πρόταση του κυρίου Πρέντα και υποστηρίχθηκε και από τον κύριο Γκόλνης από ό,τι είδαμε, αλλά εδώ δεν θέλουμε να συζητήσουμε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Θέλουμε να συζητήσουμε τον τρόπο εργασία αυτού του Κοινοβουλίου. Πρόκειται για μια κατεπίγουσα πρόταση η οποία υποβλήθηκε από το ΕΛΚ, δεν υπήρξε αρκετή υποστήριξη και τώρα προσπαθούν να την ε, συμπεριλάβουν στην Ολομέλεια. Νομίζω ότι ανεξάρτητα από το θέμα το οποίο συζητούμε, δεν είναι αποδεκτή η διαδικασία για την ε, αγαστή λειτουργία του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Θέτω το αίτημα λοιπόν προς ψήφιση. Ποιοι είναι υπέρ τη αλλαγή τη ημερήσια διάταξη, Παρακαλώ. Those again. Κατά. Απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε μεν, αλλά είναι σαφές. Ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Has everyone voted? Ψήφισαν όλοι. Πέρασε ψηφοφορία, συνάδελφοι. Απορρίπτεται. Δεν αλλάζει λοιπόν η ημερήσια διάταξη της Τρίτης. Περνάμε τώρα στην ημερήσια διάταξη της Τετάρτης. Η Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά, Πράσινη Αριστερά ζήτησε δήλωση από τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική για τις ε, θανατηφόρες επιθέσεις ε, ε, των ΗΠΑ κατά του νοσοκομείου στο Αφγανιστάν των γιατρών χωρίς σύνορα. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Τζίμερ για να συζητήσει και να υποβάλει το αίτημα εκ μέρους της ομάδας της. Κυρία Πρόεδρε, η ομάδα μου σύμφωνα με τον κανονισμό ζητάει συζήτηση χωρίς ψήφισμα για την θανατηφόρο επίθεση της Αμερικανικής ε, αεροπορίας στο ιατρείο των γιατρών χωρίς σύνορα στο Κουντούζ. Πρέπει να συζητηθεί ε, αύριο, 8.30 ώρα θεωρούμε εμείς, παρουσία της ε, κυρίας Μογκερίνη και προτείνω μάλιστα να μιλήσουν ε, όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες. Ε, το Σάββατο που μας πέρασε σκοτώθηκαν 12 ε, εργαζόμενοι και τουλάχιστον 7 ασθενείς μεταξύ των οποίων 3 παιδιά και είχαμε πάνω από 30 τραυματίες. Σύμφωνα με τους γιατρούς χωρίς σύνορα στις 3 Οκτωβρίου επλήγει το ιατρείο τους ε, στην ε, Κουντούζ ε, σε διαλύματα των 15 λεπτών. Το κεντρικό κτίριο του νοσοκομείου, στο οποίο βρίσκεται και η εντατική μονάδα αλλά και μια μονάδα ψυχοθεραπείας, επλήγησαν επανειλημμένα και με μεγάλη ακρίβεια. Ήδη στις 29 Σεπτεμβρίου είχαν δοθεί, είχε δοθεί το στίγμα του νοσοκομείου στην ε, Διεθνή Συμμαχία και στον Αφγανικό στρατό και στις ε, πολιτικές αρχές. Παρόλα αυτά βομβαρδίστηκε. Συμμετέχουν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο Αφγανιστάν, αλλά βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει και αναπτυξιακή βοήθεια και μάλιστα περισσότερη από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Πάρα πολλές οργανώσεις από την Ευρώπη βοηθούν, μεταξύ των οποίων και οι γιατροί χωρίς σύνορα. Γι' αυτό ζητάμε να διαρευνηθεί το περιστατικό. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος υπέρ, η κυρία Χάρμς. Υποστηρίζω εξ ονόματος της ομάδας μου το αίτημα της Γκάμπι Τσίμερ που πολύ καλά το τεκμηρίωσε. Πρέπει να θέσω εκ προημίου ότι με τα όσα αναφέρθηκαν και με τον λόγο του Προέδρου Ομπάμα που ζήτησε πλήρη διακρύβωση αυτών των φρικτών γεγονότων του Κουντούς όπως προανήγγειλε ανακουφίστηκα αλλά πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μια διεθνή συζήτηση για το τι συνέβη ιδιαίτερα επειδή στο Αφγανιστάν επειδή λέγω στο Αφγανιστάν οι εξελίξεις συνολικά είναι τρομακτικές και φοβίζουν και εμείς μέχρι σήμερα μια συζήτηση απουσιάζει ανάμεσά μας για αυτό το θέμα. Δεδομένων των συζητήσεων αύριο, δεδομένη της παγκόσμιας κατάστασης, όλα επιχειρηματολογούν υπέρ του ότι αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης για το Αφγανιστάν, λόγω των φρικτών γεγονότων του κουντούς που περιέγραψε η κυρία Τσίμερ, πρέπει να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη εργασιών μας. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος κατάφτυσης πρότασης, παρακαλώ. Αν δεν συμβαίνει αυτό, τότε θα ψηφίσουμε επί του αιτήματο. Όσοι είναι υπέρ τη αλλαγή στην ημερήσια διάταξη, να σηκώσετε τα χέρια. Όσοι είναι εναντίον. Αυτό το αίτημα έγινε δεκτό. Και έτσι τώρα θα έχουμε μια δήλωση θα ελέγξουμε συνάδελφοι, αλλά ήταν σαφές από εδώ που κάθομαι. Λοιπόν, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για αυτή την πρόταση αλλαγής της ημερήσιας διάταξης και προσθήκης. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Συνάδελφοι, έγινε δεκτό το αίτημα, είναι σαφές. Έτσι αλλάζει η ημερήσια διάταξη της Πέμπτης με αυτή την προσθήκη. Θα έχουμε μια δήλωση επ' αυτού του θέματος την Πέμπτη το πρωί και η Σύνοδος θα αρχίσει στις 8.30 οι εργασίες μας στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Ζητήσατε τον λόγο κυρία εσείς. Όχι αυστηρά για την ίδια την ημερήσια διάταξη αλλά για την τρίτη για τη συζήτηση <clears throat> για την ε, Dieselgate. Έχω αντιληφθεί ότι η διάσκεψη των Προέδρων σε σχέση με τον Αντιπρόεδρο Τίμερμανς που ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμμετάσχει σε αυτή τη συζήτηση βλέπουμε ότι η Επίτροπος Μπιενκόφσκα τώρα θα είναι παρούσα που είναι υπέρ του επιχειρήν και της ε, εσωτερικής αγοράς. Δεδομένης όμως της σοβαρότητας του θέματος και μια και αφορούν περιβαλλοντικές πολιτικές, πολιτικές ε, διαχείρισης, διακυβέρνησης και άλλα θέματα Τέσσερις κοινοβουλευτικές επιτροπές του Κοινοβουλίου εμπλέκονται σε αυτό το θέμα και θα θέλαμε να κατανοήσουμε και να αντιληφθούμε γιατί, για ποιους λόγους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ανταποκρίνεται στο αίτημά μας και δεν αποστέλει, αποστέλει τον Αντιπρόεδρο Τίμερ μας σε αυτή τη συζήτηση. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Η Επιτροπή πρέπει να αποφασίζει ποιοι θα συμμετάσχουν στη συζήτηση πάντα οι επίτροποι ομιλούν εξ ονόματο τη Επιτροπή όταν παρίστανται στην Ολομέλεια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει πρόταση για αλλαγή τη ημερήσια διάταξη περαιτέρω για την Πέμπτη. Η διάταξη των εργασιών καθορίστηκε πλέον. Υπάρχει όμω ένα διαδικαστικό. Κύριε Σμιτ, έχετε τον λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να θίξω ένα θέμα για την Τετάρτη για την ημερησία διάταξη σε σχέση με τα όσα αναφέρατε πιο πριν σε σχέση με το, ε, τις, τις εργασίες μας η ε, καταληκτική ε, προθεσμία για τις τροπολογίες θα είναι αύριο και για την κατάθεση τροπολογίες που περιορίζει σε σχέση με την, ε, με την συμμετοχή από 4 σε 3 από πλευρά του κυρίου Σούλτ χωρί κανένα λόγο κάτι τέτοιο ε, γίνεται δεκτό από ένα ηλεκτρονικό μήνυμα κάποιος από τη διοίκηση λέει ότι θα ήταν κατά της, ε, των, θεμάτων πρωτοκόλου ή εθιμοτυπίας. Δεν νομίζω ότι μια και είναι τέτοια η σημασία αυτού του θέματος ε, και μάλιστα υπάρχει και η πρόσφατη ε, τεκμηρίωση για την κατάθεση και αποδοχή τροπολογίας. Θα ήθελα λοιπόν να είναι πολύ πιο τεκμηριωμένη η ανάλυση για το τι συμβαίνει και τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει στην και την αλλαγή ημερησίας διάταξης ή εργασιών. Γιατί αν δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια ανάλυση σε βάθος, δεν είναι δυνατόν να ψηφίζουμε για θέματα των εργασιών αυτών που ίσως μετά τροποποιούνται. Ευχαριστώ. Θα γνωρίζετε κύριε ότι αυτό το θέμα στο 2014 είχε τεθεί και η ίδια τροπολογία θεωρήθηκε, τότε μη αποδεκτή με βάση την νομική ερμηνεία που δόθηκε στον πρόεδρο τότε δεν άλλαξε τίποτα από τότε και η απόφαση του πρόεδρου είναι τελεσίδικη από αυτού του θέματος και δεν είναι αποδεκτή αυτή η τροπολογία και δεν μπορούν να γίνουν άλλα σχόλια. Προ, ε, συνάδελφοι, παρακαλώ. Ο κύριος Πρέντα, έχετε διαδικαστικό κύριε Πρέντα. Ευχαριστώ πρόεδρε θα ήθελα εγώ από πλευράς μου να αναφερθώ στην κατεπίγουσα κατάσταση σε σχέση με την πέμπτη το πρωί. Είναι η δεύτερη φορά που θα έχουμε τέσσερα θέματα αντί τριών θεμάτων υποσυζήτηση. Θα ήθελα και πάλι να σας υπενθυμίσω τι αναφέρει το άρθρο 135 του κανονισμού μας του Ευρωκοινοβουλίου. Παράθεμα το, ο συνολικός αριθμός θεμάτων που μπορεί να εισαχθεί όσον αφορά τα κατεπήγοντα στην ημερήσια διάταξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία θέματα, ακόμα και με υποκεφάλαια τα οποία μπορεί να εντάσσονται. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχουμε τέσσερα τώρα θέματα. Επειδή επέμεινε ο πρόεδρος Σούλτς να προσθεθεί ένα τέταρτο θέμα και έτσι για, για δεύτερη φορά παρεύει, ε, παρεμβαίνοντας παρεύει τους κανόνες. Θα ήθελα να επανέλθουμε στα τρία θέματα όπως προβλέπει ο κανονισμός. Αν έχουμε τέσσερα θέματα, θέματα θα έχουμε λιγότερο χρόνο να συζητήσουμε. Δεν πρέπει να παραβαίνουμε τους κανόνες και κανονισμούς μας. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Πρέντα. Από ό,τι γνωρίζω υπήρχε συμφωνία στην διάσκεψη των Προεδρών επ' αυτού του θέματος και υπήρχε προφορικό έτοιμο για αλλαγή τη ημερησία διάταξη. Πολύ καλά τεκμηριώσατε τη θέση σα και την άποψή σα και θα γνωστοποιηθεί και στον πρόεδρο τη υπηρεσία. Περνάμε στο πρώτο θέμα τη ημερησία διάταξη απόψε.